Συνάδελφοι, παρακαλώ θερμά καθίστε για να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Δεν έχουμε βέβαια σήμερα τόσο πολλά σημεία όσο χθες, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να επιτελέσουμε το καθήκον μας. κάποιες ανακοινώσεις πρώτα. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης ε, έχουν μοιραστεί, υπάρχουν παρατηρήσεις, αντιρρήσεις. Όχι. Οπότε θεωρώ συγκεκριμένα τα πρακτικά. γραπτή δήλωση 2-2010 της κυρίας Μακοβέη, του κυρίου Μπουσουτήλ, Ντεμαγκίστρης, Αναγκόμες και Μπαρτ Στάς για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Η δήλωση αυτή έχει υπογραφεί από τους περισσότερους ευρωβουλευτές και η γραπτή αυτή δήλωση με βάση το άρθρο 123 θα μοιραστεί στους αποδέκτες και θα δημοσιευθεί με τα ονόματα των συνυπογραφόντων. Πρόκειται για ένα κείμενο που εγκρίθηκε στις 18 θα εγκριθεί στις 18 Μαΐου του 2010. Η κυρία Μάρκοβα για διαδικαστικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά του συναδέλφους που συνυπέγραψαν και εξέφρασαν την υποστήριξή του για την γραπτή αυτή δήλωση. Θα ήθελα επ' ευκαιρία να απευθύνω έκκληση προ το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να θεσπίσουν έναν ισχυρό μηχανισμό πάταξης τη διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλό τα κράτη-μέλη να δηλώσουν τη βούλησή του να πατάξουν τη διαφθορά πριν είναι πολύ αργά. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε την πρώτη έκθεση, που είναι η έκθεση του κυρίου Μέντες Δεβίγκο, ως προς την απόφαση να μην συγκληθεί συνέλευση για τη μεταρρύθμιση των συνθηκών σε ό,τι αφορά τα μεταβατικά μέτρα για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ψηφίσουμε με